Pan przewodniczący. E, kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο θέμα στην ημερησία μα διάταξη είναι η ανακοίνωση πλευρά τη Βαρόνη Άστον, η δηλώση μάλλον τη Βαρόνη Άστον για το κράτο δικαίου στη Ρωσία. Εκ μέρου τη είπα τη εκπροσώπου, παρακαλώ την κυρία Γκιόρη να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, μετά από αίτημα της Βαρόνης Άστον, η Ουγγρική Προεδρία, η οποία εκπροσωπεί, με συγχωρείτε την τη εκπρόσωπο, αντιπρόεδρο της Επιτροπής, θα ε, κάνω την εξής δήλωση. Όπως ξέρετε, η Βαρόνη Άστον ταξιδεύει στην Βόρειο Αφρική και την Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα. Θα ήθελα να θίξω το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη Ρωσία, διότι παρά τα θετικά μηνύματα του ε, Προέδρου Μετβέντεφ πέρσι, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στο Βόρειο Κάυκασο. Δυστυχώς υπάρχει βία, όκληση και εκφοβισμός κατά ακτιβιστών δικηγόρων και ανεξαρτήτων δημοσιογράφων, κάτι το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Ο αριθμός τέτοιων περιπτώσεων είναι ανησυχητικά υψηλός. Οι Ρώσοι δημοσιογράφοι Όλε Κάσιν και Ανατολή Αντάμτσουκ, καθώς και ο ακτιβιστής Κωνσταντίν Φετίσοφ, αποτελούν τις τελευταίες υπενθυμίσεις του κλίματος ανασφάλειας και εκφοβισμού κατά δημοσιογράφων στην καθημερινή τους εργασία. Παρά τις εγγύσεις από τα υψηλότερα επίπεδα, οι δράστες αυτοί δυστυχώς δεν προσάγονται στη δικαιοσύνη και δεν καταδικάσονται. Θα ήθελα να αναφέρω τις περιπτώσεις των κυρίων Εστεμίροβα, Πολιτκόφσκα, Μπαμπούροβα και Μαρκέλοφ Πρόκειται για μια μεγάλη δοκιμή και δοκιμασία για την ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος της ε, Ρωσίας. Δυστυχώς η ατιμορρησία επικρατεί. Υπάρχουν όμως και θετικές εξελίξεις. Θα πρέπει να αναφέρω εδώ την απόφαση των δημοτικών αρχών της ε, Μόσχας που επέτρεψε τις ειρηνικές διαδηλώσεις που είχαν απογορευτεί πέρσι, όπως το άρθρο 31 ή την ημέρα της οργής. Χαιρόμαστε για αυτή την απόφαση, όμως ε, ε, λαμβάνουμε στοιχεία για αφαίρετες ε, φυλακίσεις και συλλήψεις ειρηνικών διαδηλατών κατά την διάρκεια αυτών των διαδηλώσεων που είχαν επιτραπεί. Αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα. Η ελευθερία λόγου, η ελευθερία του συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε αποτελούν πρόκριμα για την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών. Όλες αυτές οι ελευθερίες έχουν κατοχυρωθεί από το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επίσης γνωρίζουμε ότι τα έχει δεχτεί η Ρωσία ε, στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει την Ρωσία να αρκεστεί σε αυτές τις υποχρεώσεις. Ο πρόεδρος Μετβέντεφ ζήτησε από το Προεδρικό Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εξετάσει τις υποθέσεις Κοντορκόφσκι-Λεμπέντεφ και Μαγνίτσκι Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την απόφαση και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αναφερθεί στη σοβαρότητα των υποθέσεων αυτών. Ο πρόεδρος Μετβέντεφ μίλησε συχνά για τον νόμιμο μηδενισμό που επικρατεί στη ε, Ρωσία. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί αρχίζοντας με την αναθεώρηση και μεταρρύθμιση του δικαιοδοτικού συστήματος στη Ρωσία. Επειδή λοιπόν θα πρέπει να ισχύσει το κράτος δικαίου, θέσαμε αυτό τον όρο ε, σαν πρόκριμα για τις εταιρικέ μας σχέσεις, για την εταιρικότητα ως προς τον εξυγχρονισμό. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ε, ένα σύστημα, την θέσπιση ενός αναιρετικού συστήματος για περιπτώσεις ποινικού και αστικού δικαίου μέσα στα πλαίσια της αντιμετώπισης της διαφθοράς και των συμβάσεων της Χάγης. Η κατάσταση στο Βόρειο Κάφκασο είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και θα πρέπει να αναλυφθεί άμεσα δράση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός Κλοπόνιν να, ότι θα πρέπει να αναλάβει μια νέα στρατηγική οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Θα πρέπει όμως να αντιμετωπιστούν και οι τρομοκράτες που πλήττουν τον αστικό πληθυσμό. Επίσης, η συνεχιζόμενη ατιμορρησία και ασυλία των, των ομάδων ασφαλείας που δρούν στην Τσετσενία είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν πρέπει να υπόκεινται αυτή τη βία άνθρωποι οι οποίοι προασπίζουν τα επαγγέλματά τους ή την κοσμοθεωρία τους. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η κατάσταση αυτή δεν ήταν και ιδιαίτερα θετική. Όμως υπάρχουν θετικά μηνύματα ως προς τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και παλινοδίες και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει επιτευχθεί μία συνολική βελτίωση. Όμως δεν πρέπει να αποθαρρυνθούμε. Ο σημαντικός αριθμός νομολογίας του ΕΔΑΔ δείχνει ότι υπάρχουν κίνητρα έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στη Ρωσία σε σχέση με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ρωσία το δέχτηκε αυτό και δέχτηκε και τις επικρίσεις εν μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε σε αυτή μας την πορεία διότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Σας ευχαριστούμε πολύ. κυρία Προεδρεύουσα και τώρα επιτρέψτε μου να στραφώ προς τις πολιτικές ομάδες για να ακούσουμε τους ομιλητές τους εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Γιώργης Σέπφλιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Είναι γνωστό ότι δεν ε, ε, ικανοποιεί τους όρους του κράτους δικαίου το σύστημα, το καθεστώς στη Ρωσία, ούτε για το διεθνές δίκαιο, ούτε για τα δικαιώματα των πολιτών τους. Έτσι λοιπόν, όταν, ε, όταν διαπραγματεύεται με τη Ρωσία η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια σειρά από παράγοντες, την πολιτική παρέμβαση, τη διαφθορά και την, τις εξάρσεις βίας. Έτσι λοιπόν ε, αβεβαιότητα αλλά και απόλυτη απουσία διαφάνειας και λογοδοσίας χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για δε τον πολίτη της Ρωσίας αυτός επηρεάζεται ακόμη περισσότερο από την ευθερεσία και τη βία και δεν ε, βλέπει πουθενά την τηρήση των ε, δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σεβασμό των οικουμενικών δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη λύση παρά να μείνουμε εμείς στη δική μας εσωτερική ε, υποτιθέμενη νομιμότητα και την ανομία που επικρατεί στη Ρωσία. Κύριο Σεβερίν, Πρόεδρο, ε, το μοντέλο διαχωρισμού τη εξουσία ανάμεσα στην κυβέρνηση και την κοινωνία. Πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικών αποφάσεων. Η προβλεψιμότητα τη διαδικασία λήψη αποφάσεων και η σωστή υλοποίηση των αποφάσεων όμως ε, ε, κατοχυρώνονται από την ειλικρίνεια, τον επαγγελματισμό και την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία μπορούν να συνεργαστούν μόνο εάν σε αυτά τα πρότυπα άσκηση εξουσίας διασφαλίσουν ότι είναι συμβατά τα δικαστικά συστήματά του. Για να υπάρξει συμβατότητα ε, θα χρειαστεί συνεργασία και εταιρική σχέση, αμοιβαία εμπιστοσύνη, διαλειτουργικότητα ε, και όχι ε, κατακρίσεις και αερολογίες. Η Ρωσία έχει υπογράψει τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Οπότε το Δικαστήριο στο Στρασβούργο είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να βασιστεί στο Συμβούλιο Ευρώπη, ώστε από κοινού με τη Ρωσία να δημιουργήσει τον ενιαίο χώρο ασφάλεια και δικαιοσύνη. Επιπροσθέτω, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει προ την προσχώρηση στη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ω νομική οντότητα, ακριβώ γι' αυτό θα πρέπει να επισπεύσει την σύγκληση και τη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα τη Ρωσία για να επικρατήσει η δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Πριν από χρόνια, κυρίε και κύριοι, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε περισσο... λίγη περισσότερη εξουσία από μία ενεργό μη κυβερνητική οργάνωση. Θυμάστε την κατάσταση και σήμερα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, όμω έχουν αλλάξει τα πράγματα και είμαστε ένα ισχυρό θεσμικό όργανο και άρα έχουμε και μεγαλύτερε ευθύνε και πρέπει να αυτοπεριοριστούμε να υπάρχει αυτοσυγκράτηση. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε ε, συναισθηματικά, δεν μπορούμε να αφήνουμε να δεκυβεύονται οι αρχέ μα. Ε, οφείλουμε να επιδιώκουμε την δίωξη και την επιβολή δικαιοσύνη και να να μην υποκύπτουμε ε, στις ε, πιέσεις ε, που ασκούν τα διάφορα λόμπι. Χρειαζόμαστε μία ενιαία προσέγγιση, αλλά και ανοιχτό πνεύμα και αυστηρότητα. Όλα αυτά θα πρέπει να καθοδηγούν τη συζήτησή μας, το διάλογό μας με τη Ρωσία, ούτω ώστε να εκπονήσουμε μία στρατηγική εταιρική σχέση και ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Η κυρία Κριστίνα Ογιούλαντ ε, από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι η Ρωσία είναι πάρα πολύ σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, ε, περιμένουμε από τη Ρωσία να τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να υλοποιεί να προστατεύει τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών τη. Ε, είναι αναμφισβήτη αλήθεια ότι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου και των βασικών ελευθεριών ε, είναι μια κοινοτυπία γιατί η Ρωσία. Είναι εκτεταμένη η διαφθορά και ε, έτσι 300.000 Ρώσοι πολίτε αποχώρησαν μόνο το 2010 από τη Ρωσία. Αυτό είναι επιβλαβέ φυσικά για όλου και είναι δύσκολο να αναπτυχθεί επιχειρηματικό πνεύμα ζούμε υπό αυτέ τι συνθήκε. Η τάξη, η δημόσια τάξη είναι αντισυγματική. Ένα από το παράδειγμα είναι η κατάσταση στο, Βόρειο, στο Νότιο Κάφκασο. Ε, και προβλέπεται πολυκομματικό σύστημα μεν στη Ρωσία, αλλά στην ουσία είναι μόνο κομματικό ε, και ε, υπάρχει μόνο ένα αγγυλωμένο κοινοβούλιο. Ζητούμε λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα και οι κυρώσει πρέπει να εφαρμοστούν κατά των Ρώσων αξιωματούχων που ευθύνονται άμεσα για τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι του κράτου δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει στην πολιτική τη ενώπιον τρίτων χωρών να δείχνει συνέπεια. Θα απαξιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αν εθελοτυφλούμε ενώ παρακολουθούμε σοβαρέ παραβιάσει δικαιωμάτων σε πολλέ χώρε, ενώ σε άλλε επιβάλλουμε κυρώσει για σε αξιόπινε πράξεις. Ε, χρειαζόμαστε συγκεκριμένε βελτιώσει στην κατάσταση στη Ρωσία. Πρέπει να δούμε κατάματα την αλήθεια. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριος Βέρνερ Σούλτς, παρακαλώ, έχουμε στον Πρασίνο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, παρά ένα πολύ καλό σύνταγμα, η Ρωσική Ομοσπονδία δεν, είναι, δεν αποτελεί κράτος δικαίου. Δεν υπάρχουν ακόμη οι βασικές προδιαγραφές για ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ελεύθερη τυπία. Το ανεξάρτητο ρωσικό δικαστήριο είναι αυτό του Στρασβούργου, λένε κάποιοι ηρωνικά. Οι Ρώσοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στα δικαστήριά τους και ξέρουν ότι δεν αποδίδεται εκεί η δικαιοσύνη. Και αυτό το δείχνουν και τα πολύ ψηλά ποσοστά εφέσεων που ασκούνται. Είναι πολύ αυτοί ε, που ε, καλούν σε εξουδετερώση του νομικού μηδενισμού ή του δικαστικού μηδενισμού που επιβάλλεται, που όμως τελικά σημαίνει ότι μόνο τη δική του ασφάλεια και επιβίωση εξυπηρετεί το καθεστώς. Αυτό βλέπουμε από την υπόθεση Ροντοκόφσκι με την επαναλαμβανόμενη καταδίκη του Ροντοκόφσκι βλέπουμε ότι το ρωσικό κράτος δεν έχει ξεπεράσει την περίοδο των Κούλακ. την ε, δίωξη των αλλοφρονούντων από το καθεστώς με όργανο τη δικαιοσύνη και με πολιτική καθοδήγηση και επιλογές σε, σε ε, α, κοινές δικαστικές διαδικασίες. Έχουμε επίσης την υπόθεση Μαγνίτσκι, ενός δικηγόρου ο οποίος θέλησε να αποκαλύψει περιπτώσεις διαφθοράς, ο οποίος συνελήφθη και ο οποίος με αποτρόπαια ιατρικά μέσα έχασε μέσα στη φυλακή τη ζωή του. Βλέπουμε ότι η τήρηση των σταγματικώς κατοχυρωμένων πολιτικών ελευθεριών δεν εξασφαλίζεται στη Ρωσία, δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις της από το διεθνές δικαίο, δεν λειτουργεί ανεξάρτητα η Ντούμα και οι προεδρικές εκλογές, δεν υπάρχει ελεύθερη θέσπιση και λειτουργία κομμάτων, δεν υπάρχει δυνατότητα για ελεύθερα μέσα μαζικοϊκής ενημέρωσης ή για ανεξάρτητη αντιπολίτευση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τσουαλ Στάνοκ, μεταρρυθμιστής όπως ξέρετε, η Ρωσία είναι ένας μεγάλος εταίρος για εμάς, αλλά δυστυχώς δεν επικρατεί το κράτος δικαίου. Δυστυχώς είχαμε να κάνουμε με ένα μη ανεξάρτητο δικαιοδοτικό σώμα, όπου καταδικάστηκαν πολλοί δημοσιογράφοι και ακτιβιστές. Βεβαίως το Κρεμλίνο θα ήθελε να νομιμοποιηθεί η κυβέρνησή της, όπως φάνηκε και γιατί, ε, όπως ξέρουμε από τα Wikileaks, δυστυχώς η Ρωσία θεωρείται ένα κράτος μαφία. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας φυσιχασμός ως προς την κατάσταση. Το ΕΔΑΔ έχει 27.000 υποθέσεις που εκκρεμούν κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και όπως ξέρετε, βλέπουμε ότι είναι παράλογο να συμμετέχει η Ρωσία στο Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ρωσία δυστυχώς αγνοεί το διεθνές δίκαιο. Πιστεύουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ξανασκεφτεί το κατά πόσο θα είναι σκόπιμο να συμμετέχει σε αυτή την οργάνωση. Αγαπητέ συνάδελφοι, συνάδελφε, μιλήσατε σχετικά γρήγορα και οι διερμηνείς αντιμετώπισαν ε, πρόβλημα, ένα σχετικό πρόβλημα. Ο κύριος Μπρούνο Πόσο καιρό έχω στη διάθεσή μου. Ένα λεπτό, εντάξει το Κοινοβούλιο θέλει να δώσει μαθήματα στη Ρωσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος ε, Τάνοκ μίλησε για τον Ζουλιάν Ασάνς, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του Wikileaks του οποίου δεν συμμερίνομαι τις δράσεις. Κρατείται εδώ και εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο για γελίους λόγους πριν εκδοθεί στη Σουηδία, πριν βεβαίως εκδοθεί και στις ΗΠΑ. Υποτίθεται ότι βίασε δύο κορίτσια, η οποία είπε, η μία είπε ότι έσπασε το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια της ε, πράξης. Και η δεύτερη είπε ότι πρόκειται για μία πράξη που έγινε με τη συνένεσή της. Εάν δεν ήθελαν να πιαστούν αυτές οι δύο κοπέλες από τον κύριο Ασάνς, δεν θα έπρεπε να μπουν γυμνές στο κρεβάτι του βλέπουμε αυτό το παράδειγμα και, και βλέπουμε, μα μιλάμε για τη Ρωσία λέει ο πρόεδρος, μην ξεφεύγουμε συνάδελφε. Μιλάμε για το θέμα της Ρωσίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Γκόλνης ε, μιλά εκτός μικροφώνου, με κλειστό το μικρόφωνο. Yeah. Dear colleague, dear Κατανοώ, συνάδελφε, αλλά στην ημερήσια διάταξη συζητάμε για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Λυπάμαι που έπρεπε να σας ε, διακόψω. Δεν πρέπει να αλλάζουμε το θέμα μας. Λυπάμαι που σας αφαίρεσα το λόγο. Τώρα, η κυρία Όμεν Ράιτεν. Για ένα λεπτό. Ναι, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση προκύπτει λόγω των πράξεων της ρωσικής ηγεσίας, με πρώτο τον κύριο Μετβέντεφ, που ισχυρίζονται ότι έχουν εξυγχρονίσει το κράτος δικαίου, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι είναι πολύ άριθμα τα συγκεκριμένα παραδείγματα της παρεμπόδισης αυτού του εξυγχρονισμού. Και κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε ότι η διαφθορά διονγκώνεται διαρκώς από ό,τι λένε ε, πηγές αξιόπιστες παρά ένα νέο νόμο κατά της διαφθοράς και ότι είναι διαρκή η παραβιάση των δικαιωμάτων. Εάν θέλουμε λοιπόν με σοβαρότητα να επιδιώξουμε τον εξυγχρονισμό κύριε Πρόεδρε, αυτό σημαίνει ότι προχωρούμε με αποτελεσματικά μέτρα. Αυτό ισχύει και για τη Ρωσία λοιπόν. Εάν η Ρωσία θέλει να μιλήσει για εξυγχρονισμό, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να έχει σχέσεις με μια εξυγχρονισμένη Ρωσία, δεν αντιλαμβάνομαι πόσο σε ένα έγγραφο για την εταιρική σχέση ο εξυγχρονισμός βρίσκει μόνο 5-6 αράδες για να εκφραστεί. Πρόεδρε, χρειαζόμαστε πολύ πιο αυστηρή και προσεκτική μελέτη της κατάστασης. Άλλωστε στο πλαίσιο της εκθέσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ρωσία θα επανέλθουμε στην αρχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλέκνιστον για δύο λεπτά. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, λυπούμε που ε, μπήκε στην εμερή διάταξη το θέμα αυτό τόσο βραχυπρόθεσμα και έτσι η πατήκ πρόσωπος δεν μπόρεσε να παραστεί στη συζήτηση. Η Κάθριν Άρστον στους τελευταίους ε, μήνες ε, συνεργάστηκε με το Συμβούλιο για μια εσωτερική διαβούλευση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια συνεργασία ε, και για τη βελτίωση των σχέσεων με τους στρατηγικούς μας εταίρους όπως η Ρωσία. Μια στονισμένη λοιπόν θέση δική μας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θα καθιστούσε απαραίτητη την παρουσία και της κυρίας Άστον στη συζήτηση αυτή η Ρωσία και γεωγραφικά αλλά και για λόγους των ιστορικών μας, του ιστορικού μας παρελθόντος έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για, για την εξέλιξη εσωτερικά της Ρωσίας, στην εσωτερική πολιτική και βέβαια ο συντονισμός των δράσεων για τον εξυγχρονισμό θα πρέπει να παρακολουθούνται από κοινού. Αυτό το κοινό πρόγραμμα εργασίας για τον εξυγχρονισμό περιλαμβάνει σημαντικές και ορθές προσεγγίσεις για την ουσιαστική υποστήριξη των εξελίξεων του κράτους, της ανάπτυξης του κράτους δικαίου στη Ρωσία. Αποτελούν ε, δηλαδή αυτές οι προσπάθειες τον ουσιαστικό τρόπο να αξιοποιήσουμε αυτήν την εταιρική σχέση προς όφελος των πολιτών. Μια πρωτοβουλία για τον εξεχωρισμό της Ρωσίας σημαίνει ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει τη δυνατότητα για επικοδομητική συνεργασία, προσφέρει μάλλον τη δυνατότητα για επικοδομητική συνεργασία και στους διεθνείς του εταίρους. Ας την αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία. Εάν θέλουμε να είναι α, βιώσιμος αυτός ο εξυγχρονισμός λοιπόν, δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στην επιδίωξη ενός τεχνολογικού εξυγχρονισμού. Τεχνολογικά εξελιγμένη κοινωνία σημαίνει ότι είναι και μια κοινωνία η οποία στηρίζεται σε ορθές αρχές δικαίου, στο κράτος δικαίου. Όταν ε, ξεφεύγει από το πλαίσιο του κράτους δικαίου μια κοινωνία δεν μπορεί να έχει το κουράγιο να προχωρήσει στην καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη. Ας βοηθήσουμε λοιπόν την Ρωσία να αγγίξει αυτόν τον εξυγχρονισμό που προσωποθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο για ένα λεπτό ο κύριος Γιάτσεκ Προτασέβιτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, πολλοί τους προλαλήσαντες, και εγώ προσυπογράφω αυτή την προφανή διαπίστωση ότι η Ρωσία είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και από γεωπολιτική άποψη και άποψη διεθνούς ασφάλειας αλλά και από οικονομική άποψη στρατηγικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν μας εκπλήσει καθόλου αυτό το ζωηρό ενδιαφέρον για την κατάσταση στη γειτονική χώρα. Υπάρχουν μερικά ανησυχητικά φαινόμενα και τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μόνο 3% των Ρώσων πιστεύει ότι ασκεί κάποια επιρροή στην πολιτικό βίο της χώρας και 60% πιστεύει ότι δεν μπορεί να προσπίσει αποτελεσματικά τα δικαίωμα ενώ το 82% των Ρώσων πιστεύει ότι δεν τηρούνται στη Ρωσία τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι πραγματικά μια θλιβερή εικόνα της κατάστασης μιας χώρας ε, που μας είναι ιδιαίτερα προσφυλής. Η οικονομική ανάπτυξη, ο εξυγχρονισμός της οικονομίας ε, ε, δεν θα πρέπει να είναι το μοναδικό στοιχείο τη συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή, όπω το κάνουμε για τι άλλε γειτονικέ μα χώρε και εταίρους. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριο Μάικλ Γκάλερ. Ευχαριστώ στα πολωνικά ο κύριος Γκάλε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκτός από την ευρύτατη συνεργασία, όχι μόνο την οικονομική, αλλά και τη συνολική στις προκλήσεις παγκοσμιοποίησης, είναι σημαντικό και φάνηκε σήμερα και ακούστηκε να δούμε την κατάσταση του κράτους δικαίου στη Ρωσία και να το διατηρούμε στην ημερησία διάταξη. Τις τελευταίες εβδομάδες μιλήσαμε πάρα πολύ για σταθερότητα και στη Μεσόγειο και ορίσαμε τι δεν είναι σταθερότητα. Οι αυταρχικές δομές δεν είναι σταθερότητα. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι και για τη Ρωσία, ε, αν δεν σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αν δεν σταματήσει η πολιτική επιρροή στη δικαιοσύνη, στα δικαστήρια, αν δεν σταματήσουν οι διώξει των δημοσιογράφων και των αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν θα πάει καλά η κατάσταση. Για μένα λοιπόν ε, πάντα είναι ε, επίκαιρο αυτό το θέμα να το συζητούμε και στις ε, σχέσεις που έχουμε ε, με τη Ρωσία και στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να το θέτουμε. Να ξεκαθαρίσουμε προς τη Ρωσία ότι διακυβεύει το ίδιο της στο μέλλον εάν δεν εξασφαλίζει το κράτος δικαίου στην επικράτειά της. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, um, Σας ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία του Catch the κύριος Κέλαμ. Είχαμε ε, δεκάδες ακτιβιστών και δημοσιογράφων που έχασαν τη ζωή τους στην Ρωσία. Πολικόφσκα, Μπεστεμίροβα, Βλατκεύσκη. Μόνο ένα, ούτε ένα έγκλημα δεν έχει διαλευκανθεί μέχρι στιγμής από αυτά και ούτε ένας δολοφόνος δεν έχει προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε λοιπόν να διαφορούμε γιατί θα, θα κριθούμε ως σε αυτά τα εγκλήματα αν δείξουμε διαφορή. Και χθε είχαμε μια περίπτωση στη διάρκεια τη ε, Χοντορκόφσκι κάποιος που δήλωσε ότι η δικαστική απόφαση έχει επιβληθεί εκ των άνω. Και τα μέτρα στην υπόθεση Μαγκρίτσκι είναι μια απόδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μας ενδιαφέρει πραγματικά η διαφάνεια και το κράτος δικαίου στην Ρωσία. Το γεγονός ότι ε, έχουν εκνευριστεί οι Ρώσοι ότι αφορά και μόνο την ιδέα μιας ε, απαγόρευσης ε, χορήγησης θεωρήσεων δείχνει πόσο σημαντική είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επέλθουν κάποιες αλλαγές στην παρούσα κατάσταση. Ο κύριος Γουότσον. Πολλοί από εμά, ε, κυρία Πρόεδρε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε τη Ρωσία ω ε, μέλο τη μεγάλη οικογένεια των ευρωπαϊκών ε, λαών. Και ελπίζαμε μετά την κατάρρευση του τείχου του Βερολίνου να έρθει η Ρωσία όλο και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που δυστυχώ δεν έγινε, γιατί η παρούσα ρωσική ηγεσία ακολούθησε το δικό τη μονοπάτι και προκάλεσε δυστυχώ απογοήτευση σε αυτού που επιδιώκαμε και επιζητούσαμε κράτο δικαίου, δημοκρατία ε, και διαφάνεια στη Ρωσία. Είχαμε πολλή εμπειρία σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τη Ρωσία και ο καθένας έχει τις δικές του εμπειρίες και βιώματα. Ελπίζουμε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πιέσει την υπατεκπρόσωπο να υιοθετήσει μια νέα πολιτική απέναντι σε οποιαδήποτε χώρα για τις οποίες καταστρατηγούν ε, περίτρανα τις ε, αξίες και αρχές που μας είναι προσφυλή. Μα ενδιαφέρει το εμπόριο, αλλά θα πρέπει να τολμήσουμε να συζητήσουμε με τη Ρωσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και Ας μην επιτρέψουμε στους ηγέτες της να ε, ξεπλένουν χρήματα στις ευρωπαϊκές τράπεζες, ε, να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους ε, στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ή να, παραθερίζουν στα ευρωπαϊκά θέατρα, θέρετρα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να, συμβαδί, να βαδίσουμε προς μια πραγματικά διοντολογική και ηθική εξωτερική πολιτική. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που λέγουν ότι χρειαζόμαστε ευφυή μέτρα για να αντιμετωπίζουμε αυταρχικά καθεστώτα τα οποία παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τους εκπροσώπους εδώ σήμερα της ΥΠΑ της εκπροσώπου να μας απαντήσουν αν είναι πρόθυμοι να λάβουν μέτρα ε, κατά εκείνων που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως ορίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, αν δεν απατώ με τις 15 Δεκεμβρίου ήταν, που ε, ζητάει πάγωμα των υπηρεσιών και απαγόρευση θεώρησης ε, διαβατηρίων 60 υπευθύνων ε, που ενέχονται στην υπόθεση Μπατμίτσκι, ο οποίο δυστυχώ έχασε τη ζωή του στη φυλακή. Δεν θα βρεθούν ένα δύο θαραλέοι υπουργοί εξωτερικών να δώσουν συνέχεια σε αυτή την υπόθεση και την πρωτοβουλία. Και οι εκπρόσωποι εδώ τη ΥΠΑ, εκπροσώπου, μπορούν να μα πούν εάν αποδειχθεί ότι εκτελούσε εντολές της κεντρικής κυβέρνησης ε, ο δικαστής που εξέδωσε την απόφαση για την υπόθεση Κοδορκόφσκη δεν θα πρέπει να προσθεθεί στη λίστα αυτή. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ρωσία είναι από τους σημαντικότερους εταίρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημοκρατική της παράδοση δεν είναι μακρά. Ε, είναι ακόμα σε διαδικασία εκδημοκρατισμού η χώρα έχει να αντιμετωπίσει και τον Ισλαμικό κίνδυνο και την Ισλαμική τρομοκρατία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικότερη εκεί η θέση των δυνάμεων ασφαλείας. Οι προδιαγραφές λοιπόν και τα πρότυπα στη Ρωσία είναι διαφορετικές από τις δικές μας. Η κατάσταση είναι πολύ ευαίσθητη και θα πρέπει να ελέγχεται πάρα πολύ προσεκτικά. Ο διάλογος με τη Ρωσία πρέπει να είναι αντικειμενικός ε, σε συνθήκες εταιρικής σχέσης βελτίωση του συστήματος ναι, αλλά θα πρέπει να μαθαίνουμε κι εμείς από τη Ρωσία να έχουμε εταιρικέ σχέσεις φιλίας, όχι να προσπαθούμε πάντα να τους δίνουμε μαθήματα. Έχουμε κοινά συμφέροντα για σταθερότητα και ειρήνη στην Ευρώπη. Thank you. Ε, in my opinion, Mr. κατά τη ε, συνέταξε ένα θεμελιωμένο και τεκμηριωμένο ψήφισμα με σωστά συμπεράσματα. Αλλά ίσως ε, δεν κατάλαβα το επιχείρημα του κυρίου Φλέκενστάιν. Γιατί αν ε, οι διαδικαστικοί κανόνες δεν μου επιτρέπουν να θέσω μια ερώτηση, τον ερωτώ. Τι πιστεύει δηλαδή, θα πρέπει να απόσχουμε ε, στην ε, ψηφοφορία του ψηφίσματος ή αντίθετα τάχθηκε υπέρ της αμέρης υποστήριξης των σοσιαλιστών προς το ψήφισμα. Γιατί δεν κατάλαβα. Κύριε Φλέκενστάιν, θα θέλετε να απαντήσετε. I didn't listen. Sorry. But I, but I come back to you Θα ήθελα να δώσω την ευαίσθηση στον κύριο Τάραντ να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Παρακαλώ κύριε Τάραντ. Κοιτάξτε, δεν είμαι σίγουρος ε, κατά πόσον ε, προτείνεται να υποστηρίξουμε αυτό το ψήφισμα ή κατά πόσον μας καλείτε να απέχουμε σε αυτή την ολομέλεια, να δηλώσουμε αποχή. I will vote for the... Ε, εγώ θα έλεγα να ψηφίσουμε υπέρ. Μάλιστα, ωραία. Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία Catch the Eye. Οπότε θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της είπε της εκπροσώπου στην Προεδρεύουσα της Ουγγρικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς, Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω όλους για τις εύστοχες ερωτήσεις που θέσατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Κατανοώ πολύ τα μελήματά σας, μελήματα που εκφράσατε πολύ και ανησυχίε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να τα θέτει υπόψη αυτά σε όλα τα επίπεδα στου Ρώσου συνομιλητέ μα. Δεν θα πρέπει να διστάσουμε ε, να θέτουμε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα και ερωτήματα. Εάν θέλουμε να δρούμε ω στρατηγική εταίρη, και εγώ πιστεύω ότι είμαι θα στρατηγική εταίρη της Ρωσίας, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουμε και θέματα καθόδη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι Χάρηκα ιδιαίτερα για δύο λόγους κατά τη διάρκεια της παρούς συζήτησης. Ο πρώτο είναι ότι κανείς δεν αμφισβήτησε ότι η Ρωσία είναι σημαντικός εταιρικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο, ήταν γενική η συμφωνία ε, στο ημικύκλιο ότι ο εξχρονισμός και η σταθεροποίηση μιας πλήρους δημοκρατίας και του κράτους δικαίου δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί στη Ρωσία. Ε, παραμένουν πολλά προβλήματα με τις ε, λειτουργίες και της δημοκρατίας στη Ρωσία. Οπωσδήποτε θα διαβιβάσω όλα τα θέματα που θίξατε στην ύπατη εκπρόσωπο και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να δώσουμε συνέχεια και να παρακολουθήσουμε διάφορους τρόπους τα θέματα αυτά τους τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας. Η επικείμενη επίσκεψη της ρωσικής κυβέρνησης της Βρυξέλλης 21 ε, του μηνός Φεβρουαρίου θα μας δώσει πολύ ε, μεγάλη ευκαιρία και δυνατότητα να θέσουμε αυτά τα ζητήματα. Οφείλω εδώ να προσθέσω ότι η Ρωσία είναι μόνιμο και διαρκές θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και πρέπει να γνωρίζετε και ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, συζήτησε πρόσφατα τα θέματα αυτά της αδίκων σχέσεων με τη Ρωσία. Πέρσι το Σεπτέμβριο συγκεκριμένα και πιστεύω ότι ο πρόεδρος Παν ε, Ρόμπαϊ θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Επιτρέψτε μου να απαντήσω αμέσως σε κάποια μέλη που έθεσαν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτος, στην κυρία Χάουταλα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είπατε εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ε, πολύ σοβαρά υπόψη. Το ψήφισμα που εγκρίνεται τον περασμένο Δεκέμβριο. Σε ό,τι αφορά το Σεργέη Μακνίσκι και τη Βέρα Κρυφόνοβα, ε, θα πρέπει να διερευνηθούν σε βάθο αυτέ οι υποθέσει και βεβαίω το Συμβούλιο ε, Εξωτερικών Υποθέσεων που αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Εξακολουθούμε να θέτουμε αυτή την ανησυχία και το μέλημα υπόψη των Ρώσων σε όλα τα επίπεδα, ε, όχι ε, μόνο στις τακτικές επαφές που έχουμε, αλλά και σε επίπεδο συνόδων κορυφής. Οποιαδήποτε απόφαση για περιοριστικά μέτρα θα εξεταστεί από το Συμβούλιο, αλλά θα πρέπει να γίνεται χρήση προσεκτική αυτών των ε, μέσων, έχοντας γνώση της υπόθεσης και μετά από διερεύνηση. Θα απαντήσω στην κυρία Όμεν Ρόιτε να μου επιτρέπετε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πραγματικά στον πυρήνα των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία και θα τα θέσουμε υπόψη των Ρώσων σε πολλά επίπεδα. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας, ιδιαίτερα και τα δικαιώματα προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Στην ε, παρούσα συμφωνία, στη μελλοντική μάλλον συμφωνία, είναι πολύ βασικό στοιχείο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να συνοψίσω ε, κάτι που είπα προηγουμένως η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κράτος δικαιού θα πρέπει να παραμένουν αναπόσπαστα τμήματα των προσπαθειών εξυγχρονισμού που ε, διεξάγονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πρόθυμη να υποστηρίζει τη Ρωσία στις προσπάθειες αυτές. Η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία του συνέρχεστε, και του συνεταιρίζεστε ε, είναι ε, πραγματικά ε, πάρα πολύ βασικά στοιχεία για όλες τις δυτικές δημοκρατίες. Θα πρέπει να επαναλάβει τις νομικές της δεσμεύσεις η Ρωσία και να, τις, να ανταποκριθεί σε αυτές. Έχει αναλάβει υποχρεώσεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στα Ηνωμένα Έθνη και στον ΟΑΣΕ. Παραμένει ζήτημα βαθιάς ανησυχίας για μας ο Βόρειος Κάφκασος. Θα πρέπει να εθαρρύνουμε τη Ρωσία να ζητήσει αηφόρο και βιώσιμη λύση σε αυτό το ενδυμικό πρόβλημα της περιοχή. Το σημαντικό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές ανησυχίες, αλλά έχει και πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει η Ρωσία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και θετικέ εξελίξει. Θα πρέπει να πιστέψουμε τον πρόεδρο Μετβέντεφ και να συνεχίσουμε το σοβαρό διάλογο με τη Ρωσία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα αν υπάρχουν υποθέσεις θα πρέπει να τις παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και να τις γνωρίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύτιμα σχόλιά σας και είπα ότι εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ενημερωθεί δεόντως για τις απόψεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε κυρία Γκέρι. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 12 σήμερα το μεσημέρι. Α, συγγνώμη, διορθώνει η πρόεδρος. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη το μεσημέρι στις 12. Διακοπή μέχρι το μεσημέρι στις 12.